τους για τη διαχείριση των αλλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Ε, διαδικαστικό. Α, για το Catch the Eye, μάλιστα. Η κυρία Ούλρικε Ρόντου στη συγγετρία, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Έχουμε μία έκθεση ιδέας πρωτοβουλίας για να θέσουμε ένα ερώτημα, να φέρουμε κάτι ή να θέσουμε στο επίκεντρο κάποιε συγκεκριμένε περιφέρειε. Εδώ μιλάμε για τη διαχείριση των αλληλευτικών στόχων στι εξόχω απόκεντρε περιοχέ. Αυτό είναι ο στόχο ε, τη έκθεση, ε, να αναπτυχθούν καλύτερα ε, στοιχεία για τα προγράμματα, ιδίω σε ό,τι αφορά και τα αποθέματα, την κατάσταση των αποθεμάτων. Επίση, θέλουμε να μειώσουμε την άναρχη παράνομη αδήλωτη αλία. Θέλουμε λοιπόν να ληφθούν ενεργά μέτρα παρακολούθησης και διαπραγμάτευσης με τις γειτονικές χώρες με τις οποίες ε, δεν έχουν ε, υπογραφεί συνθήκες, ε, μάλλον ληφτικές συμφωνίες. Θέλουμε να λάβουμε υπόψη και να προασπίσουμε τα συμφέροντα των ληφτικών στόχων των εξόχων ε, περιοχών διότι υπάρχουν θέσεις εργασίας που προσφέρει ο αλληλευτικός τομέας ε, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό για την αλία ε, και για τις εξόχους από κεντρές περιοχές. Θα πρέπει να κάνουμε σχετικές επαληθεύσεις. Θέλουμε να δούμε την ένταση των ενισχύσεων. Παραδείγματος χάρη θέλουμε να αυξήσουμε την ενίσχυση για την αντικατάσταση κινητήρων των σκαφών. Πρέπει να πω ότι ήδη υπάρχει ε, πρόβλεψη για καλύτερη επιδότηση για 100% συγκεκριμένα ε, σε, αυτούς τους, ε, σε, αυτούς τους, σε αυτές τις χώρες. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα την ένταση των ενισχύσεων σε άλλους τομείς έχει ανέβει στο 35%. θα πρέπει να αξιοποιούνται κατά το μέγιστο δυνατό οι διάφορες διατάξεις, γενικές και ειδικέ και θα πρέπει να αξιοποιηθούν καλύτερα και τα ε, ερευνητικά και επενδυτικά, ερευνητικές και επενδυτικές δυνατότητες. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις που προβλέπουν ουσιαστικά υπονοούν μια εξαίρεση, μια παρέκκληση. Αυτό έρχεται να ε, ε, ως προσθήκη. Θα πρέπει να το δούμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, ε, τροπολογίες, σε ό,τι αφορά και τις δημόσιες ενισχύσεις στην Επιτροπή Αλίας, υπάρχει η συγκεκριμένη τροπολογία, αλλά δεν έγινε δεκτή και επανέρχεται τώρα στην Ολομέλεια σε ό,τι αφορά τις αλλιευτικές ικανότητες. θα πρέπει να πω σε σχέση με αυτή την τροπολογία ότι η αντικατάσταση μεταξύ παλαιού και νέου είναι κάτι το οποίο ε, επιτρέπεται και σήμερα. Το θέμα είναι τι γίνεται με τη χρήση των ε, των δημόσιων κονδυλίων. Βάση είναι το 349 της συνθήκης ε, που πράγματι μπορεί να είναι η βάση για ειδικά μέτρα στον ε, ε, το Μετσαλία εξόγως από τις περιφέρειες, αλλά αυτά τα ειδικά μέτρα θα πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο ώστε να υπάρχει συνεκτικότητα, να μην υπονομεύεται συνεκτικότητα της κοινής ελευτικής πολιτικής. Η κοινή ελευτική πολιτική Έχουμε και το ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και λες δεν επιτρέπει δημόσια χρηματοδότηση για ανανέωση του στόλου. Και έχουμε και το άρθρο 11 του πολίτες που πρέπει να λυθεί υπόψη. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν φιλοπεριβαλλοντικές αλλιευτικές ε, πρακτικές. Ε, θα πρέπει να δούμε τα αντίστοιχα άρθρα. Θέλουμε να υπάρχει ε, συνεκτικότητα, γι' αυτό και δεν θεωρούμε ότι είναι συνάδει με τις διατάξεις και τις πρακτικές η δημόσια επιδότηση και ενίσχυση. Γι' αυτό λοιπόν θα καταψηφίσω τη σχετική τροπολογία, διότι είναι και κατά της κανσελευτικής πολιτικής και ανήκει το κουτί της Πανδώρας. Και βέβαια, ε, πολύ δικαιολογημένα, εάν γίνει αυτό για τις εξώξεις από τις περιφέρειες, θα το διεκδικήσουν και άλλες περιοχές στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Επίτροπος Έτιγκερ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και την εισηγήτρια συγκεκριμένα την κυρία Λουρίκη Ρόντου αλλά και την ομάδα της ε, για την ε, πολύ αντικειμενική ε, έκθεση αυτή της πρωτοβουλίας. Δεν είμαι η Δήμον, διάβασα την έκθεση και κατάλαβα κάποια πράγματα. Νομίζω ότι είναι άρτια, εξετάζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αλληλευτικός τομέας ε, σε αυτές τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Αναφέρονται πολύ συγκεκριμένα μέτρα τα οποία προτείνονται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και για τη σταθεροποίηση του τομέα. Εμείς ε, δεχόμαστε και ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης δραστηριοποιούμαστε από αυτού, δηλαδή σε ό,τι αφορά τις εξόχως απόκεντρες ε, περιοχές να βρούμε λύσεις ε, για τα προβλήματα και ε, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της κοινής πολιτικής και στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Ήδη δε έχουμε, πιστεύω, ήδη κάνει πολύ σημαντικά βήματα και ατενίζοντας προς το μέλλον. Θα δούμε και στον επόμενο προπολογισμό. και στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού ακόμη περισσότερο ε, πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε στις συστάσεις σας και στις προτάσεις σας αυτά τα μέτρα και ε, να τα βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο. Μιλάμε για κάποιες, ε, κάποια τήματα πληστικής πρόσβασης, μέτρα για μικρούς, μικρής κλίμακας στόλους και μεγαλύτερη ένταση των ενισχύσεων. Μερικά είναι μόνο αυτά από τα μέτρα τα οποία αναφέρεται στη δική σας την έκθεση. Φυσικά θα πρέπει να παρακολουθήσουμε και να πλησιώσουμε τους ε, περιφερειακούς, ε, εθνικούς και τοπικούς ε, οργανισμούς στο, έργο τους, ε, διότι δεν αρκεί το ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει και οι περιφερειακές και εθνικές αρχές να συμμετέχουν. Είναι πάρα πολύ σημαντική, ιδίω στον τομέα αυτό, οι οργανισμοί στο περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και οι αρχές. Προτείνουμε ένα νέο πλάσιο στη για τις ε, εξόγως κεντρές ε, περιοχές. Βέβαια, τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία έχουν ε, την ευθύνη, όπως και τα ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και οι επιχειρηματίες από τον κλάδο της αλίας. Εγώ νομίζω πάντως ότι αυτή η είναι μια πολύ καλή βάση, την οποία εμείς λαμβάνουμε υπόψη και οι αρμόδιοι ε, συνεργάτες μας ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβουν υπόψη ε, την έκθεση της κυρίας Ρόντους και είμαστε στη διάθεση και της κυρίας Ρόντους προσωπικά και όλων ημών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους τώρα της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, το λόγο κύριο Σαμαρζέ. De quelle surpêche? Υπεραλίευση. Ε, ποιοι είναι ένοχοι στον Ινδικό ωκεανό από όπου έρχομαι, οι κάτοικοι της Ρεϊνιό αλλιεύουν το 0,16%. Ε, 0,16% του συνόλου των αλλιευμάτων, 250 τόνους όλους και όλους, από το 1.600.000 τόνους που αλλιεύονται από τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς στόλους. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια βαθύτατη αδικία. Και ακριβώς αυτό θέλει να διορθώσει η τροπολογία μας. Αυτό το οποίο προτείνουμε είναι λογικό. Ξέρετε ότι θα πρέπει να σεβόμεθα πλήρως την αηφορία στον τομέα της αλίας. Άλλωστε η έκθεση της Επιτροπής Ρέγγι έκανε την ίδια πρόταση. Αύριο λοιπόν πέραν των, α, της ψευδολογίας και εν πλήρη γαλήνη Ας στηρίξουμε τις ε, ε, ακραία περιφερειακές ε, ζώνες γιατί κινδυνεύουν να καταστραφούν. Ευχαριστώ. κυρία Μοντέρα Αγκιάρ έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Για μία ακόμη φορά βλέπουμε σήμερα πόσο σημαντική είναι η γαλάζια οικονομία τα ναυτιλιακά ζητήματα, αλλά η σημασία κυρίω τη αλίας για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Ε, ζητώ τη συμβολή όλων τοπικών και περιφερειακών παραγόντων και των πολιτικών εθνών για να καθορίσουμε μια πραγματικά κοινή αλληλευτική πολιτική. Σήμερα βλέπουμε ότι μα χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό όργανο που θα αφορά την Αλία, όπως ισχύει και για τη γεωργία. Θέλουμε μια πιο αλληλέγγυη Ευρώπη, μια πιο κοινωνική Ευρώπη, μια Ευρώπη που θα σέβεται και θα τηρεί τις συνθήκες της. Δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε στη μοίρα του τους, εξω, τους, τους των εξόχως απόκεντρων περιοχών, γιατί και αυτή είναι πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να στηρίξουμε την ανανέωση του αλληλευτικού στόχου των από απόκεντρων περιοχών. Αυτό δεν δεκυβεύει ούτε το Ταμείο Θάλασσα και Αλίας, ούτε την κοινή αλληλευτική πολιτική. Απλώς εξασφαλίζει την υγεία όσων εργάζονται ε, στη θάλασσα και συμβάλλει στην καλύτερη διατήρηση των αλληλευτικών πόρων. Ελπίζω όλες οι πολιτικές ομάδες να συμφωνήσουν για αυτό το θέμα και έτσι νομίζω ότι δεν θα απογοητεύσουμε τους ε, πολίτες που μας εξέλεξαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκ μέρους ε, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, το λόγο κύριο Σεράου Σάντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω ε, την κυρία Ρόντουστ για το έργο και την αφοσίωσή της. Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές έχουν ε, μεγάλες διαφορές από τις υπόλοιπες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξού και το ειδικό άρθρο που προβλέπει η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτό το νομικό πλαίσιο, η έκθεση πρωτοβουλίας πολύ σωστά απευθύνει έκκληση για τη δημιουργία ενός ε, χρηματοδοτικού μέσου που θα ευνοεί αυτές τις περιοχές για να χορηγούνται ε, δημόσιες ενισχύσει στις περιοχές αυτές για την αντικατάσταση των αλληλευτικών του πόρων, αύριο θα ψηφίσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό να μπορούν οι σε αυτών των από απόκεντρο περιοχών να λαμβάνουν δημόσιες ενισχύσει κάτι που δεν θίγει είναι την κοινή αλληλευτική πολιτική. Απλώς απαιτεί μια τροποποίηση της σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί ε, η παροχή δημοσίων ενισχύσεων για την ανέωση του ελευτικού στόρου τη ΕΑΠ δεν αντιβαίνει ούτε έχει παρεμποδιστεί από την κοινή πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική αλλά από την σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πέρασε χωρίς καμία διαβούλευση με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Τόμασιτς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει φυσικά να αφιερώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όλες τις πολιτικέ και ε, γιατί πραγματικά είναι απομονωμένες και γεωγραφικά και για άλλους λόγους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αντίστοιχη προσοχή θα πρέπει να δείξουμε για παρόμοια προβλήματα που έχουν νησιωτικές περιοχές και σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στην Κροατία, γιατί η μοίρα των αλλιέων της Κροατίας από στα κροατικά νησιά είναι ίδια με αυτή και των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Γι' αυτό ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει τη σχετική ε, οδηγία για τη Μεσόγειο, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα ελευτικά τους μέσα ή κάτοικοι των μεσογειακών νησιών για την άσκηση της ε, παράκτιας αλίας. Και μάλιστα θα ήθελα να υποστηρίξω την, ε, την έκθεση αυτή και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που πέρυσι υποστήριξαν την δική μου έκθεση για το θέμα αυτό. Η κυρία Μπαραντίκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση για το καθεστώ ε, του ελευτικού στόχου στι εξόχω απόκεντρε περιοχέ είναι μια μοναδική ευκαιρία καταπληκτική για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να περάσει από τα λόγια στα έργα και να ζητήσει συνοχή, ενσυναίσθηση και κατανόηση ε, από τις οργανώσεις που κατά παράδοση και εσφαλμένα ε, συνδέουν τις ελευτικές ικανότητες με την προσβολή των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Οι, Ευρωπαίοι αλληλείς είναι αυτοί που έχουν συμφέρον για την ε, βιωσιμότητα των ελευτικών πόρων. Το άκουσα με τα αυτιά μου από τους αλληλείς από τα Κανάρια. Γι' αυτό και χωρίς επιφυλάξεις θα στηρίξω το δικαίωμά τους σε κοινοτικέ ενισχύσεις για να ανανεώσουν τους τόλους τους. Έτσι θα βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και ε, υγείας σε ένα ε, περιβάλλον που χρειάζεται καλύτερη και περισσότερη απασχόληση. Μιλούμε για πιο ενεργειακά αποδοτικά σκάφη, θα ρηπαίνουν λιγότερο και θα ε, είναι πιο σύγχρονα. Ε, δεν ζητούμε αύξηση τη ελευτική ικανότητα, γιατί η βελτίωση του ελευτικού στόχου δεν γίνεται ει βάρο τη διατάραξη ισορροπία μεταξύ αλίευση και διατήρηση. Επίση, θα ήθελα να σα παροτρύνω να εκπονήσετε μια σοβαρή μελέτη για τον αντίκτυπο Τη αερασιτεχνικής αλίας στις ζώνες αυτέ. Αυτό με ζητά ο ελευτικό κλάδο σε περιοχέ που ε, αυξάνεται ο τουρισμό. Γιατί οι επαγγελματίε του κλάδου έχουν δικαίωμα και ζητούν περισσότερε πληροφορίε και έλεγχο αυτή τη ερασιτεχνική αλίας που λόγω των διαστάσεων που έχει λάβει επηρεάζει και ασκεί πιέσει στη διαχείριση των αλληλευτικών πόρων. Σα ευχαριστώ. 1,5 λεπτό ακριβώ Μπράβο σα. Εκ μέρου τη ε, ΓΚΟΕ, ο κύριο Φερέιρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση αναγνωρίζει ότι η κοινή ελευτική πολιτική δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των εξόχων απόκεντρων περιοχών. Είναι ένα θετικό βήμα που απαιτεί, όμως, τουλάχιστον κάποιες ε, νομοθετικές ε, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις των κακών κειμένων. Θέλουμε ε, ζητούμε την πρόταση ενός, ζητούμε την δημιουργία ενός νέου ΠΟΣΕ για την αλία για να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες και να καταπολεμήσουμε τα μειονεκτήματα αυτών των περιοχών. Ε, φυσικά χρειάζεται εξυγχρονισμός και ανανέωση του ελευτικού στόλου των ε, εξόχως απόκεντρων περιοχών. Γι' αυτό ε, είμαστε υπέρ της έκθεσης που είναι ισορροπημένη και πολύ σωστή. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε μάχη υπέρ της διεύρυνσης των ζωνών αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ε, και επίσης ε, τη διεύρυνση από τα 100 στα 200 ναυτικά μίλια. Και θα, θα ταχθούμε υπέρ ε, μέσω θετικής διάκρισης για παράκτια μικρής κλίμακας αλίας προκειμένου να διατηρηθεί η περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο αλλιευτικός στόλος έχει αρχίσει και είναι πλέον ε, μεγάλης ηλικία 30 με 40 ετών. Δυστυχώς και τα αλλιεύματα μειώνονται. Υπάρχει λαθροαλία επίσης. τα χρήματα που δίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη δεν επιτρέπουν την ανανέωση δυστυχώς του των μικρών αλλιευτικών σκαφών. Οι απαγορεύσεις δυστυχώς συνεχίζουν να σοβούν χωρίς αμφισβήτηση. Θυμίζω ότι στις περιοχές της υπερπόντιες της Γαλλίας υπάρχει τεράστια ανεργία των νέων και η αλληλεία θα μπορούσε να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης σε αυτά τα ξεχασμένα εδάφη, διευκολύνοντας και την αηφορία στην αλία. Μάτο. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η έκθεση αυτή και για την περιοχή των Καναρίων. Γενικά είναι ένα ουσιαστικό μέσο για τις απομεμακρυσμένες περιφέρειες Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες ε, για την αλληλεία στις περιοχές αυτές που θα δώσουν ευκαιρίες στους νέους να απασχοληθούν. Ένα σημείο το οποίο πρέπει να μας ε, απασχολήσει είναι η αυστηρή τήρηση των κανόνων για την αηφορία στην αλληλεία θα πρέπει οι αλληλείς αυτών των περιοχών να μπορούν να αλλιεύουν και όχι να χάνουν τα αλλιεύματά τους από άλλους. Ε, δεν είναι δυνατόν να ανταγωνιστούν τους διεθνείς στόλους η τοπικοί στολείς και οι αλλιευτικοί όταν ε, έχουν στη διάθεσή τους πολύ περιορισμένα και ξεπερασμένα τεχνικά μέσα. Εμείς δεν ζητάμε ε, για να δώσουμε περισσότερα χρήματα για την ανανέωση του στόλου χωρίς κανένα όριο. Θέλουμε απλά ε, να δώσουμε κάποιες ευκαιρίες στις, στους αλληλείς των περιοχών αυτών. Δεν θέλουμε πλέον δημαγωγία, θέλουμε να μην ε, λαμβάνονται μέτρα εις βάρος των περιοχών αυτών Αυτά τα οποία προτείνει σε ορισμένα σημεία η έκθεση είναι σαφώς αβέβαια. Κυρία Τόμα, παρακαλώ. Merci, Monsieur le Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Συνάδελφοι, οι απότερες περιφέρειες της Ένωσης αντιμετωπίζουν σοβαρή κρίση και ε, πολλές φορές οι δυνατότητες οι αλλιευτικές ε, πολλούνται και οι ποσοστώσεις που υπάρχουν δίδονται σε τρίτες χώρες. Λόγω της πολύ μεγάλης απόστασης οι περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Τα, η εξαίρεση η οποία υπάρχει για την ανανέωση του στόλου ε, είναι απαραίτητη γιατί τα σκάφη είναι και περιορισμένου μεγέθους αλλά και ξεπερασμένα τεχνικά. Πρέπει να επιτρέψουμε στους αλλοιείς να αλλιεύουν με σωστό τρόπο. Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα τα περιβαλλοντικά στις ε, τροπολογίες τις οποίες προτείνουμε. Δεν προτείνουμε την αύξηση των ποσοστώσεων. Ε, είμαστε υπέρ της αηφορίας, απλά πρέπει να αντικατασταθούν τα ξεπερασμένα σκάφη από νέα ε, και αποδότικα. Ας μην υποκύπτουμε στην παραπληροφόρηση. Ευχαριστώ. Περνάμε στο Catch the Eye. Ο κύριος Βέρνερ Κούν είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, με επίτροπε. Μπορώ να ε, στηρίξω απόλυτα αυτά που είπε η σας σε μια συζήτηση ε, ανεξαρτήτως του για ποιον τομέα μιλάμε. Ε, εδώ μιλάμε για την αλληλεία. Το θέμα είναι ε, ε, η η κλίμακα της ενίσχυσης στους πιο μικρούς φορείς. Εδώ τώρα μπορούμε ε, και πρέπει να δραστηριοποιηθούμε χωρίς να δαπανίσουμε πάρα πολλά χρήματα με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Νομίζω ότι μπορούμε κάτι να κάνουμε. Θέλουμε την ανακαίνιση, τον εξυγχρονισμό, ε, αλλά μιλάμε για πολύ μικρής κλίμακας, ε, πολύ μικρού μεγέθους στόλους ε, πώς μπορούν αυτοί οι αλληλείς ε, να ψαρέψουν. Μιλήσαμε για την Ρενών, για τη Γουαδελούπη, για τέτοιες εξόχως απόκεντρες ε, περιφέρειες, όπου ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός με αλληλείς από την υπηρετική Ευρώπη. Δεν καταλαβαίνω όλο αυτό το πρόβλημα. Λέγεται πολύ ξεκάθαρα και στην τροπολογία ότι θα πρέπει να τα ελέγξει η Κομισιόν και να δει κατά πόσον είναι δυνατή αυτή η χρηματοδότηση για αυτά τα μικρά παραδοσιακά λιευτικά σκάφη και βέβαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εθνικοί πόροι, όχι μόνο Και Το θέμα είναι να δώσουμε ένα μήνυμα ε, στη μικρή παραδοσιακή αλία. Και αν θέλουμε να το κάνουμε πρέπει να υπερψηφίσουμε αυτή την ε, τροπολογία. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να στηρίξω το έργο της συναδέλφου Λρίκη Ρότου. Είμαι όμως ε, Κανάριος. Ε, είμαστε σε μια εξόχω απόκεντρη περιοχή. Εκεί ε, αναφέρονται μόνο ε, τα συγκεκριμένα ε, εδάφη που αναφέρονται στο 349 και υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που προβλέπονται και στο πρωτογενές και στο παράγωγο δίκαιο για αυτές τις περιοχές και νομίζω ότι αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει αν θέλουμε να προστατεύσουμε την μικρή κλίμακα παραδοσιακή αλλά και ερασιτεχνική αλία και στα Κανάρια νησιά για να υπάρξουν συγκεκριμένες ενισχύσεις για την ανακαίνιση ενός απαρχαιωμένου στόλου για να βελτιωθούν οι γεωνομικές συνθήκες και αλλά και συνθήκες ασφαλείας όπως επίσης και να διορθωθούν κάποια περιβαλλοντικά ζητήματα, γιατί χρησιμοποιούνται μέχρι στιγμής πιο ρηπογόνα καύσιμα που πρέπει να πάψει να και δεν θέλουμε ε, να αυξήσουμε λευτικέ δυνατότητε, γιατί σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να γίνει αυτό με αυτό το πολύ μικρή ε, κλίμακα στόλο. Απλά ε, θα δώσουμε δυνατότητε σε αυτά τα άτομα που έχουν σάρκα και οστά, που έχουν πάθο και αυτό το επάγγελμα που κάνουν, να του δώσουμε δυνατότητα να επιβιώσουν. Μιλάμε για λιγότερο ευνημένε περιοχέ, για πάρα πολύ απομακρυσμένε τι εξόδου τις περιοχέ, αυτέ θέλουμε να στηρίξουμε. Ευχαριστούμε κύριε Αγγελάρ. Ο κύριο Νότης Μαριάς παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές πρέπει πράγματι να τύχουν της προσοχής του Κοινοβουλίου μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό βέβαια μας δίνει την ευκαιρία να στραφούμε και προς τη Μεσόγειο, διότι και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και μάλιστα οι όροι του άρθρου 349 της Συνθήκης έχουν σχέση και με τα μικρά νησιά στη Μεσόγειο, ιδίως τα μικρά ελληνικά νησιά διότι εκεί υπάρχει πάλι μικρή έκταση δύσκολη μορφολογία του εδάφους οικονομική εξάρτηση από μικρό αριθμό προϊόντων και απόσταση. άρα λοιπόν και για την μεσόγειο και ιδίως για την ελλάδα πρέπει να έχουμε ρυθμίσεις σε σχέση με την οδηγία που αφορά την παράκτη αλληλεία και να έχουμε αλλαγές για να μπορούμε επιτέλους να στηρίξουμε τον εξυγχρονισμό του στόλου να έχουμε θετικά μέτρα υπέρ των αλλιέων να έχουμε ένα ειδικό καθεστώς ουσιαστικά στο πλαίσιο της κοινή αλλιευτικής πολιτικής με παρεμβάσεις κρατικές αλλά και με ενισχύσεις από πλευράς ευρωπαϊκής ένωσης. θα ήθελα ο κύριος επίτροπος ο κύριος έτιγκερ να δει και αυτό το θέμα στο μέλλον. ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ένα είναι το βασικό χαρακτηριστικό της ελευτική δραστηριότητας σε από απόκεντρες περιοχές. Ε, το χαρακτηριστικό αυτό είναι η ιδιαιτερότητα αυτών των περιοχών. Η ιδιαιτερότητα που μας καλεί να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και να λαμβάνουμε υπόψη αυτές, αυτή τη μεγάλη ιδιαιτερότητα. Είτε μιλούμε για τα νησιά του Ατλαντικού, είτε μιλούμε για τα νησιά του Ινδικού ωκεανού ε, ακόμα και μεταξύ τους διαφέρουν αυτές ε, οι εξόχως κέντρες περιοχές και φυσικά διαφέρουν ε, ριζικά από την ε, υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να μην ξεχνούμε και τα μεσογειακά νησιά που επίσης έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να επιμείνουμε στα νησιά αυτά που ζουν πολύ διαφορετικά από ότι εμείς ε, στην υπηρετική Ευρώπη. Γι' αυτό σας ζητώ να υπερψηφίσουμε την έκθεση αυτή, να ε, κρατήσουμε συνοχή ε, στην κοινή ελευθερική πολιτική, αλλά πρώτα απ' όλα να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτών των περιφερειών και περιοχών. Ο κύριος Νικολά Καπούτο, τελευταίος στη διαδικασία Κάτσε Διάη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην έκθεση την οποία καλούμεθα να ψηφίσουμε αύριο υπογραμμίζεται το ότι οι απότερες αυτές ε, γεωγραφικά περιοχές ε, θα πρέπει να μπορέσουν να ανανεώσουν τους αλλιευτικούς τους στόλους, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο και θα πρέπει να λάβουμε λοιπόν τα μέτρα και σε επίπεδο εθνικό και σε επίπεδο κοινοτικό που θα χρησιμοποιηθούν ε, για την βελτίωση και τον εξυγχρονισμό των αλλιευτικών στόλων. Έτσι θα διασφαλίσουμε και την ασφάλεια της λειτουργίας των σκαφών αλλά και ε, τον περιβαλλοντικό σεβασμό θα πρέπει και η μελλοντική ε, αλλιευτική πολιτική να λάβει υπόψη και τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν οι κλιματολογικές αλλαγές στην συγκεκριμένη αυτή ε, παράκτια ιδιαίτερα δραστηριότητα. Θα πρέπει να πάρουμε κάθε μέτρο λοιπόν έτσι ώστε ο τομέας της αλληλείας να μην ε, αντιμετωπίσει περισσότερα προβλήματα. Και για την ολοκλήρωση της συζήτησης θα δώσουμε το λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Ρόντους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Καταλαβαίνω ότι σε μερικέ εξόχω κεντρές περιφέρειε επικρατεί φτώχεια και αυτό είναι και ο λόγο ο βασικό για τον οποίο εκπονήσαμε αυτή την έκθεση. Δύο πρωτοβουλία φυσικά οι ε, συνθήκε ε, στι εξόχω κεντρές ε, περιφέρειε και ιδίω σε ό,τι αφορά την αλληλεία δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτό που ισχύει στην πυροτική Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε και τι εξαιρέσει από την κοινή αλληλευτική πολιτική και από τις άλλες διατάξει για να ληφθούν υπόψη ιδιαιτερότητε. και πρέπει να σας πω ότι έχω λάβει υπόψη μου στην έκθεση και άλλες ιδιαιτερότητε και προτείνω βελτιώσει. Εδώ επιχειρηματολογείται υπέρ τη ανακαίνησης του στόλου. Ε, λέτε ότι ε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση υπερεκμετάλλευση, στο αντίθετο, ε, πάρα πολύ χαμηλή εκμετάλλευση των αποθεμάτων αλλά μιλάτε και για την ε, ε, ρήπανση. Ε, δεν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, παραδείγματο χάρη, τη ρήπανση από τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στι φυτίες και πώς μπορεί να καταλήγουν επίσης αυτά τα υπογονωσίστε και στα νερά. Ε, το θέμα είναι να υπάρχει ε, μια ισορροπία. Σίγουρα, ε, σίγουρα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις αλληλευτικές δυνατότητες ε, και τα ηχθή αποθέματα. χρειαζόμαστε βέβαια για να κάνουμε τις σωστές αναλύσεις τα κατάλληλα στοιχεία που δεν είναι επαρκή και πρέπει ποιοτικά τουλάχιστον να βελτιωθούν. Στο μεταξύ όμως, σε ό,τι αφορά τις δημόσιες ενισχύσεις, τις, για τη χρηματοδότησή τη, της ανακαίνησης ε, του στόλου. Πού προσκοπεί και τελικά ε, έχω μια ρητορική πιο πολύ ερώτηση αυτοί οι οποίοι ε, προσυπογράφουν τροπολογία, αλλά δεν είναι από εξόχω από κέντρη περιοχή. Πώ θα εξηγήσουν στου αλληλείς από τις δικές τους περιοχές ε, για αυτή την ε, χρηματοδότηση που ζητούν για, τις, για τους των εξόχω από κέντρο περιοχή και όχι για του δικού του αλληλείς. Δεν είναι τόσο ξεχωριστή, δεν είναι τόσο ιδιαίτερη. Εγώ πραγματικά θέλω να αποφύγουμε να ανοίξουμε επαναλαμβάνω το κουτί τη Πανδώρας, ώστε και άλλοι αλληλείς εντός Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Υπηρετική ζητήσουν αντίστοιχε ενισχύσεις. Υπάρχουν ε, κάποια λύση, 30-40 ετών, που με πολύ μεγάλη χαρά θα ε, ζητήσουν επιδότηση και Γι' αυτό και θέλω να καταρριφθεί, ε, να απορριφθεί αυτή η τροπολογία. Ευχαριστώ.